να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Όταν ανέλαβα τη θέση πριν από 1,5 χρόνο του Επιτρόπου υπεύθυνου για θέματα δικαιοσύνης και ελευθερίας, ανέλαβα μία σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και συστήματα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών. SIS και VIS. Είναι μια κοινή σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και μίας σύμπραξης εταιριών. Η συμφωνία υπεγράφει το 2003. Πρόκειται για την σύνδεση ενός κεντρικού συστήματος με συστήματα εθνικά και με ειδικέ και πάρα πολύ απαιτητικέ προδιαγραφές. Προσπάθησα λοιπόν να ενημερώσω το Κοινοβούλιο από την αρχή αυτής της διαδικασίας για τις εξελίξεις και μετά τα Συμβούλια Δικαιοσύνης και Εσωτερικά θέματα τον ε, Φεβρουάριο, ενημέρωσα τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, τον Ζεχάρ Ντεπρέ, για τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με το σύστημα SIS2. Κύριε Κοέλο, έχετε λάβει αντίγραφο αυτής της ενημέρωσης, καθώς είστε συνήθως ο εισηγητής για τα θέματα αυτά και ξέρω ότι τα παρακολουθείτε πολύ στενά. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα ακριβώς επειδή με διακατέχει πνεύμα διαφάνειας, να σας δώσω πολλές πληροφορίες. Όλα τα μεγάλα βιομηχανικά προγράμματα, έτσι και το SIS και το VIS, περιέχουν ε, δυνατότητες να ξεπεραστούν οι προθεσμίες και να ξεπεραστεί και ο προϋπολογισμός. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι ικανοποιητική όσον αφορά το SIS 2 ούτε και το ΒΙΣ από αυτή την άποψη. Και παρόλο που υπήρξε κινητοποίηση και των κρατών μελών και των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλα αυτά το SIS 2 συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες και εμπόδια και το ΒΙΣ, το δεύτερο πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει μια φάση πολύ σημαντική. Οι αρχικές προδιαγραφές δημιούργησαν δυσκολίες όσον αφορά τις πρώτες δοκιμές. Φαίνεται όμως ότι σύμφωνα με την τελευταία απόφαση των κρατών μελών, η αναθεώρηση των προδιαγραφών των αρχικών θα επιτρέψουν στις δοκιμές να συνεχιστούν. Όσον αφορά το SIS-2, η σύμπραξη των εταιριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κρατη έχει ξεκινήσει την ε, προετοιμασία των προδιαγραφών μετά από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα στις 4 και 5 Ιουνίου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στη φάση της τεχνικής προετοιμασίας μιας δοκιμής που λέγεται τεχνικό όριο ή ορόσημο, milestone, έτσι ώστε να βασιστεί η φάση αυτή του προγράμματος σε υγιείς βάσεις. Η Επιτροπή έχει διαπραγματευτεί με τη σύμπραξη εταιριών όσον αφορά τις συμβατικές απαιτήσει. Γι' αυτό το πρώτο ορόσημο, τεχνικό ορόσημο. Το ποσό που χρειάζεται είναι 1.026.000 ευρώ. Ενδυναμώσαμε τη διακυβέρνηση του προγράμματος αυτού καθώς και τις συμβατικές κυρώσεις έτσι ώστε να αυξήσουμε την πίεση επί των εταιριών. Την Παρασκευή το βράδυ συνάντησα τον Γενικό Διευθυντή υπεύθυνο του προγράμματος και του ζήτησα να με ενημερώσει προσωπικά για το τι είναι τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν αναλυφθεί για να ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες. Όπως είχαμε προβλέψει τον Ιούνιο στο Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε και τις προετοιμασίες για να υπάρξει ενδεχομένως επιλογή του εναλλακτικού σεναρίου εάν αποτύχει η παρούσα τεχνική λύση. Για να λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα και το νέο χρονοδιάγραμμα θα χρειαστεί όλη αυτή η πραγματικότητα να μεταφερθεί και στο νομοθετικό επίπεδο. Γι' αυτό προτείναμε τροπολογίες για το SIS 2 με διαδικασία διαβούλευσης και του κοινοβουλίου σας για τις τροπολογίες αυτές έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να εξετάσουμε λεπτομερώς το όλο θέμα. Τώρα, για το ΒΙΣ. Σε επίπεδο κεντρικού συστήματος, τον Απρίλιο του 2009, ο ανάδοχος έκανε μία σειρά από δοκιμές που ήταν αναγκαίες για να αξιολογηθούν οι πρόοδοι που είχαν σημειωθεί. Ο ανάδοχος δεν έχει ωστόσο ακόμα καταφέρει να καλύψει όλα τα τις συμβατικές προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η σειρά των δοκιμών. Και παρόλο που του δόθηκε μια συμπληρωματική προθεσμία, δεν κατάφερε, όπως σας είπα, να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες αυτές τις δοκιμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε τη διαδικασία των συμβατικών κυρώσεων για να τιμωρηθεί ο ανάδοχος για αυτή την καθυστέρηση και τον προειδοποίησε για όλα τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν. Δεν νομίζω, αλλά ίσως διαψευστώ, ότι υπάρχει πρόβλημα σχεδιασμού. Φαίνεται ότι το STT προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς. 11 Νοεμβρίου αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές. Παράλληλα όμως τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τα δικά τους εθνικά συστήματα για να χρησιμοποιούν το ΒΙΣ. Τρία τουλάχιστον όμως κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε αυτό το τομέα. Και οι καθυστερήσεις που προέρχονται από αυτά τα τρία κράτη-μέλη είναι πιο σημαντικές από τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο κεντρικού συστήματος. Αυτή λοιπόν τη στιγμή με τα κράτη-μέλη από κοινού προβαίνουμε σε μια ενδελεχή ανάλυση προκειμένου να ορίσουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα για το ξεκίνημα του ΒΙΣ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σαφή εικόνα για την ολοκλήρωση των δοκιμών του κεντρικού συστήματος. Η συνάντηση που είχα την περασμένη Παρασκευή μου επέτρεψε να πιστέψω ότι 11 Νοεμβρίου θα είναι η στιγμή που θα ξέρουμε αν οι δοκιμές που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή χώρα θα είναι ή όχι θετικές. Εν πάση περιπτώσει όμως στα εθνικά συστήματα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά τα, τα εθνικά συστήματα για να τεθεί σε, εκείνη για να λειτουργήσει και το κεντρικό σύστημα. Ολοκληρώνω λοιπόν, μακρηγόρησα και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ήθελα να σας αναφέρω λεπτομερώς πού βρίσκονται, σε ποιο στάδιο έχουν φτάσει τα δύο προγράμματα ΣΥΣ2 και ΒΙΣ. Υπάρχουν ανησυχίες οι οποίες είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Δεν σας το κρύβω. Η τεχνική, πολιτική και δημοσιονομική κίνδυνη που υπάρχουν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να επαγρυπνούμε και να κινητοποιηθούμε διότι έχουν κινητοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί καθόλου αμεληταία κονδύλια. Το συνολικό ποσό των ε, δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κομισιόν για το SIS2 ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια πάνω σε αυτό το ποσό, πάνω από το ίμιση, 44,5 εκατομμύρια έχουν ήδη ε, διατεθεί μέχρι σήμερα. Το συνολικό ποσό για το ΒΙΣ ανέρχεται σήμερα σε 74 74 μισό εκατομμύρια. 43 εκατομμύρια έχουν ήδη δαπανηθεί μέχρι σήμερα. Αυτά τα ποσά είναι αντίστοιχα εκείνων που έχουν διατεθεί στην Ευρώπη και αλλού για ανάλογα προγράμματα τέτοιας εμβέλειας. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να ενημερώνω τακτικά το Κοινοβούλιο για όλες τις εξελίξεις που θα έχουν πιθανώς επιπτώσεις στον προϋπολογισμό ή στην ημερομηνία παράδοσης αυτών των συστημάτων. Εάν πετύχουμε με το SAS2 και το VIS θα έχουμε προσφέρει στην Ευρώπη το πιο αποδοτικό, το πιο αποτελεσματικό σύστημα στον κόσμο. Γι' αυτό με ψυχραιμία, διάβια και ρεαλισμό πρέπει να ξεπεράσουμε τυχόν εμπόδια που θα προκύψουν και ζητώ σε αυτό τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. την οποία χρειάζομαι για να παρακολουθούμε από κοντά αυτές τις δύο υποθέσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν επιτυχώς. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Θα ήθελα καταρχήν, εξ ονόματος των ε, πολιτικών ομάδων, να δώσω το λόγο ε, για το ΕΛΚ στον κύριο Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώντας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Αντιπρόεδρο Μπαρό για τις εξηγήσει του. Και θα ήθελα και εγώ να εξηγήσω γιατί θέλαμε να γίνει αυτή η συζήτηση. Θέλαμε και το ζητήσαμε γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή για την περιοχή Σέγγεν, στην οποία υπάρχει η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών. Παρόλο λοιπόν που θέλουμε να υπάρχει αυτή η πλήρης ελευθερία, δεν θέλουμε, επουδενή λόγο, να υπάρχει και ελεύθερη εγκληματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς και αυτό το σύστημα SIS θα περάσει στην δεύτερη γενιά SIS 2 ενισχύοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την ίδια ώρα περιορίζοντας την οποιαδήποτε ελευθερία για τους εγκληματίες. Πρόκειται για ένα σύστημα νέας γενιάς, το SIS-2, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε βέβαια να είναι έτοιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και τα συστήματα αυτά, κατά την άποψή μας, μπορεί να έχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση στην Επιτροπή. Ποιοι είναι οι λόγοι για ε, αυτές τις καθυστερήσεις, τι εγγυήσεις έχουμε σήμερα ότι το νέο σύστημα θα μπορέσει να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί όπως περιμένουμε και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο τελικός μας στόχος που είναι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή για να υλοποιηθεί αυτό που όλοι επιθυμούμε, δηλαδή η περιοχή Σέγγεν να προστατεύει τους πολίτες και να σταματά κάθε εγκληματική πρόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο Κλοντ Μπουράς για τρία λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πραγματικά μας δώσατε πολύ χρήσιμες πληροφορίες όπως και ο κύριος Μπουζουτήλ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις πολύ σοβαρές ανησυχίες μας για αυτές τις καθυστερήσεις. Ε, περιμένουμε όλοι να περάσουμε από το ΣΥΣ στο ΣΥΣ 2. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ βάσιμη ανησυχία. Ακούσαμε και τον ε, κύριο Κοέλιο και άλλους που εδώ και πολύ καιρό εκφράζουν αυτήν την ε, δυσαρέσκεια και ανησυχία. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο θέλει να εργάζεται ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τόσο λεπτά θέματα όπως αυτά τα δεδομένα με διαφάνεια και χρειαζόμαστε σαν Κοινοβούλιο τακτική ενημέρωση. Θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε και υπάρχει σήμερα αυτή η καθυστέρηση. Δεν νομίζω ότι ζητάμε τίποτα το παράλογο. Ζητάμε πράγματα τα οποία είναι λογικά και τα οποία απλώς απαιτούν κάποιες απαντήσεις και πληροφορίες από εσά. Πρώτον, για ποιου λόγου ε, υπάρχει τέτοια καθυστέρηση. Δεύτερον, τι εγγύσει μπορείτε να μα δώσετε σήμερα ότι αυτό θα καλυφθεί στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για του πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για όλου του πολίτε που κυκλοφορούν στην περιοχή του Σέγγεν να υπάρξει διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Και πιστεύω ότι με διαφάνεια θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των καθυστερήσεων. Πρόκειται για τεχνικά θέματα και βεβαίω αυτή η κατάσταση δεν μπορεί παρά να μας κάνει να ανησυχούμε. Πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν ε, τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις στα δικά τους συστήματα και βάσεις δεδομένων. Χρειάζεται όμως εδώ εμπιστοσύνη του κοινού. Είναι ζωτική σημασίας. Γι' αυτό και όλα τα πολιτικά κόμματα και σε συνεργασία θα πρέπει να δούμε πώς προέκυψαν αυτά τα προβλήματα, με ποιον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον και πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία του παρελθόντος, να αποκομίσουμε μαθήματα και να έχουμε μια συνολική επιτήρηση του συστήματος. Χρειάζεται να ξεπεραστούν τα τεχνικά ε, προβλήματα και δυσκολίες, αλλά χρειάζεται να επανέλθουμε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Το κοινό πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτά που γίνονται, πρέπει να υπάρξει μια μελέτη και να δούμε πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η Σάρα Λάτφορτ, εξ των φιλελευθέρων, είναι η επόμενη ομιλήτρια για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ποτέ δεν είχα τόσο χρόνο αγόρευση στα δέκα χρόνια που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δέκα λεπτά συνολικά είναι μια θαυμάσια, απίστευτη πολυτέλεια, εν πάση περιπτώσει. Είμαι ευγνώμων ε, στον Αντιπρόεδρο Μπαρό για την παρουσία του και την ενημέρωση που μας έκανα για τα προβλήματα που υπάρχουν Ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε αυτή την ενημέρωση. Όσοι γνωρίζουν ε, κάτι για τα προγράμματα πληροφορικής μεγάλης εμβέλειας ε, στις χώρες τους, ε, ξέρουν ότι αυτά τα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα είναι συχνό φαινόμενο. Αλλά όταν έχουμε δύο τόσο σημαντικά μεγάλα συστήματα, το SIS2 και το σύστημα ενημέρωσης για τις θεωρήσεις που δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, δεν εξελίσσονται ομαλά. Αυτό οπωσδήποτε βλάπτει την αξιοπιστία της ε, κοινότητας και της πολιτικής των θεωρήσεων που εφαρμόζει. Βεβαίω, είμαστε υποπίεση να περάσουμε την αναγκαία νομοθεσία διότι θέλουμε να λειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό αυτά τα συστήματα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στο πρόγραμμα είναι απογοήτευση για όλους μας. Και ήθελα να ρωτήσω επίσης ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για εκείνους που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση, για βίζα. Θα υπάρξει σύγχυση σε αυτούς τους ανθρώπους όταν το σύστημα δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις αιτήσει διαθεωρήσεις και προκύπτουν ε, προβλήματα και καθυστερήσεις. Είπατε ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις στους αναδόχους βάσει της σύμβασης λόγω καθυστερήσεων στην ε, υλοποίηση του ΒΙΣ. Τι είναι αυτές οι κυρώσεις, μπορείτε να μας πείτε τι είναι το προβλεπόμενο επιπλέον κόστος και μπορείτε επίσης να μας πείτε κύριε Μπαρό εάν εξακολουθείτε να έχετε εμπιστοσύνη στον ανάδοχο. Ή υπάρχει περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης. Οπωσδήποτε όλο αυτό έχει, θα έχει επιπτώσεις και στη σύσταση της ε, αρμοδίας αρχής που θα αναλάβει τη λειτουργία των δύο συστημάτων και της βάσης δεδομένων στο μέλλον. Οι φιλοδοξίες που είχαμε για τη συλλογή των δεδομένων ίσως θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν. Αν ε, παραμένουν αυτά τα τεχνικά προβλήματα σε επίπεδο υποδομής του συστήματος. Η σημερινή εκτίμηση για το SAS2 είναι ότι θα καταστεί λειτουργικό στο τέλος του 2011. Είναι πολύ πιθανό ότι θα υπάρξουν όμως καθυστερήσεις. Το καλοκαίρι του 2012 θα λάβουν χώρα, θα εορταστούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο. Το, η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν εφάρμοσε το SIS 1 Υπήρχε η δυνατότητα αυτή, αλλά μας είπαν ότι θα περιμένουμε το SIS 2. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ανησυχίε, μα λένε, για θέματα ασφάλεια. Μπορεί λοιπόν να μην κινδυνεύσει η αγγλική η ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση εάν το σύστημα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά το 2012 όταν θα λάβουν χώρα στο Λονδίνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κύριε Μπαρό ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον τομέα της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στο Λονδίνο και επειδή είναι εκεί και η εκλογική μου περιφέρεια. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα αυτό, η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που απασχολεί ιδιαίτερα. Περιμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια για τους πράσινους είναι η Τατιάνα Ζανόπε για τρία λεπτά. thank you. I would also on behalf of... Ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, της ομάδας μου ευχαριστώ τον Επίτροπο Μπαρό για τις ε, εξηγήσεις που μας έδωσε και, και εμείς ε, λυπούμαστε πολύ για αυτές τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Αλλά θέλω να διατυπώσω και μερικές άλλες ανησυχίες η θέση της ομάδας μας είναι πολύ σαφής σε ό,τι αφορά τη χρήση βιομετρικών ε, στοιχείων και δεδομένων στα πλαίσια του ΣΥΣ 2 και του ΒΙΣ. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω με την ευκαιρία αυτή τη θέση μας και όπως και η Σάρα Λάτφορντ Είμαι πολύ ευγνώμων για τα όχι 10 αλλά τα 6 λεπτά που μου δώσατε. Σπάνια και για μένα αυτή η πολυτέλεια. Όλο και περισσότερες αρχές από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα και αυτό με ανησυχεί. Φοβούμαστε μήπως από τεχνικό εργαλείο, σύστημα εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου. Και πρέπει, πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου μας ε, την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της υιοθέτηση των αναγκαίων νομικών ε, κειμένων και μέσων που θα ε, εξασφαλίσουν την τήρηση των βασικών εγγύσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, θέλω επίσης να αναφερθώ στην έλλειψη συνεργασίας από πλευράς ε, του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά με αξιόπιστα στοιχεία για όλη την εξέλιξη του συστήματος. Δεν θέλω να επαναλάβω την ίδια ερώτηση για που ετέθη προηγουμένως για τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή και τι θα συμβεί εάν δεν ε, είναι ικανοποιητικές είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα των δοκιμών και τι είναι το κόστος, τι κόστος πάγονται όλα αυτά. Εάν από την αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει στην όλη διαδικασία θα είχαμε ε, αποφύγει πάρα πολλά από αυτά που συνέβησαν και ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα μάθημα για το μέλλον και να, υπάρξει, και να μπορούμε να υπολογίσουμε στο μέλλον συνεργασία θα είναι πολύ πιο εκτεταμένη. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των για δύο λεπτά ο Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως και εμείς έχουμε υπογράψει αυτή το κοινό κείμενο και με μεγάλη χαρά θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε εδώ την Επιτροπή. Πρόκειται για κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογούμενων και θα θέλαμε να μας δώσει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση η Επιτροπή. Βεβαίως υπάρχει εδώ θέμα προστασίας δεδομένων, ανταλλαγής απόρριτων στοιχείων. Το θέμα είναι όμως ότι τα συστήματα αυτά ακόμα δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πλέον αμφιβάλλουμε αν το πρόγραμμα είναι βιώσιμο. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσει η Επιτροπή γιατί τέτοιες σπατάλες, γιατί ξεπεράστηκαν οι προθεσμίες. Ζητάμε λοιπόν απαντήσεις, ζητάμε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και όσον αφορά τα τεχνικά και όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Όπως λέει και το κείμενο, το Ενωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλήρως μέρος του Σέγγεν, και άλλα όμως κράτη-μέλη είναι στην ίδια κατάσταση και δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το σύστημα ΣΥΣ πριν βρεθεί μια λύση. Και θα πρέπει επίσης να δει πίεση προς τις εταιρείες που ε, βρίσκονται στην σύμπραξη έτσι ώστε να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη κύρωση προς αυτές. Είναι πολύ σημαντικό τα συστήματα να λειτουργήσουν και το πρόγραμμα να προχωρήσει. Υπάρχει όμως μέλλον για τα προγράμματα αυτά ή θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή την όλη πρωτοβουλία όπως ο Επίτροπος Μπαρό μόλις μας είπε. Υπάρχουν χώρες που καθυστερούν. Δεν υπάρχει όμως εμπιστοσύνη και αυτό δικαιολογεί ίσως αυτές τις ε, καθυστερήσεις. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να ενημερωθεί για την ανάπτυξη αυτών των σχεδίων και μέχρι να μας απαντήσει η Επιτροπή τα ερωτήματά μας παραμένουν ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ. Εξ ονόματος της ε, Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Έχετε τέσσερα λεπτά. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνούμε με τις ανησυχίες του ΕΛΚ. Πιστεύουμε ότι η συνέχιση των προσπαθειών από το SIS, το SIS2, από πολιτικής απόψεως, είναι λανθασμένες. Πρόκειται εδώ για συστήματα τα οποία αναμειγνύουν απόρριτα δεδομένα, δεδομένα μυστικών υπηρεσιών, προσωπικά δεδομένα, με έναν αλεξέλεγκτο τρόπο, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο και την ίδια ώρα βλέπουμε να υπάρχουν και βιομετρικά δεδομένα και το SIS-2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς για τους οποίους αρχικά δεν προβλέπεται. Θέλουμε λοιπόν να εξεταστεί η μέχρι τώρα φάση ανάπτυξης. Έχουμε πάρα πολλές ε, κριτικές που έχουμε ήδη εκφράσει. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη με τον ίδιο τρόπο. Πολύ απλά σας λέω ότι αφού απέτυχε το SIS-2, θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια αναπροσαρμογή και νέα κατανομή των κονδυλίων, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με πιο φιδωλό τρόπο. Υπάρχουν όντως τεράστιες καθυστερήσεις στο SIS2, αλλά επαναλαμβάνω ότι στην Γερμανία, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία και την Πολωνία, ξέρουμε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως τα κονδύλια αυτά για άλλους σκοπούς, για μια σταθεροποίηση κατάστασης και όχι για τέτοια προγράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κοέλιο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Μπαρόσο για τη δήλωσή του. Θα ήταν όμως καλό να ακούσουμε και την ε, θέση του Συμβουλίου γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούμε να ελέγξουμε πολύ καλύτερο Κοινοβούλιο την Κομισιόν αλλά όχι το Συμβούλιο. Εμείς δώσαμε εντολή στην Κομισιόν να εκτελέσει το δεύτερο ΣΥΣ το οποίο έπρεπε να αρχίσει να δουλεύει τον Μάιο του 2007. Και δεν δουλεύει όμως το σύστημα για ορισμένου, δεν θα δουλέψει μέχρι το 2012 και κάποιοι άλλοι το αμφισβητούν το ίδιο το σχέδιο. Και πέρα από το πρόβλημα του ΣΥΣ υπάρχει το πρόβλημα του ΒΙΣ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που η ίδια εταιρεία ε, έχει εκπονήσει. Πάντως, ε, εγώ θέλω να συγχαρώ τον ε, κύριο Μπαρό για όλη την προσπάθεια που κάνει, η οποία διέπεται από έντονα ευρωπαϊστικό πνεύμα. Το ΣΥΣ δεν το ξεκίνησε ο κύριος Μπαρό, το κληρονόμησε. Όταν ανέλαβε τον τομέα αυτό κατόπιν ετήματος του κυρίου Μπαρόσο. Το Κοινοβούλιο είναι αρχή του προϋπολογισμού και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν. Με το ΣΥΣ 2 εμείς θέλουμε να ελέγχουμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα, να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουν προβλεφθεί δύο milestone, ένα τον Δεκέμβριο, δηλαδή δύο τεστ, ένα τον Δεκέμβριο και το άλλο το καλοκαίρι του 2010. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την αξιόπιστη λειτουργία του ΣΥΣΕ 2 για 22 ώρες ώστε να αποδειχτεί ότι όλο το κεντρικό σύστημα δουλεύει επαρκώς. Ερωτήσεις όμως. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να εμποδίσει το τεστ που έχει προβλεφθεί. Προβλέπετε να μειώσετε τον αριθμό των χωρών που θα συμμετέχουν στην άσκηση ή σκοπεύετε να μειώσετε τα ζητούμενα τα οποία προβάλλετε. Θα ζητήσετε περισσότερα στοιχεία μετά από τα τεστ θα αυξήσετε τις απαιτήσεις σας και πόσα θα διαχειριστείτε τις ανάγκες που θα προκύψουν σε οικονομικό επίπεδο. Στο παρελθόν όταν τα τεστ δεν πήγαν καλά η εταιρεία πλήρωσε πρόστιμα. Έχει προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο και με αυτήν την εταιρεία και σε περίπτωση που έχουμε switch off υπάρχει περίπτωση να αποζημιώσει αυτή η εταιρεία. Αληθεύει τώρα ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν θέλουν να μπουν στο ΣΥΣ 2 και θα παραμείνουν στο ΣΥΣ 1. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα παρόλα αυτά να παραμείνουμε στο χρόνο ομιλίας, παρόλο που μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάσερα. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο ομιλίας. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαστε υπέρ των πρόσφατων ε, προτάσεων. Εγώ έχω πραγματικά ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θέλω να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, θεωρώ ότι το χρειαζόμαστε επιγόντως, ιδιαίτερα για τα νέα κράτη-μέλη, για να μπορούσαν να λειτουργήσουν τα συστήματα. Τα νέα κράτη-μέλη χρειάζονται αυτό το σύστημα. Αυτή λοιπόν η καθυστέρηση, η χρονική καθυστέρηση, θα πρέπει να αναλυθεί σωστά και θα πρέπει επίσης να υπάρξουν συνέπειες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την μέχρι τώρα εμπειρία για να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις στο μέλλον. Θα ήθελα να πιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο και δεν έχει νόημα εδώ να προτείνουμε τεράστιους συμβιβασμούς στη σύμπραξη εταιριών. Αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι αποτελεσματική χρήση των συστημάτων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τις ε, εμπλεκόμενες εταιρείες με οικονομικές κυρώσεις έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη σύνδεση με τα συστήματα των κρατών μέλων, διαφάνεια και μία σαφή αντιμετώπιση προς όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αναλάβει το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό από μέρους της Επιτροπής αλλά και από μέρους όλων των εταιριών έτσι ώστε να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις κάτι που θα αποφύγει περαιτέρω καθυστερήσει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Edith Bauer έχει δύο λεπτά, είναι επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για τα νέα κράτη-μέλη λέγοντας ότι θα πρέπει και εμείς βάσει του κεκτημένου του για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Χρειαζόμαστε όμως το σύστημα ΣΥΣ2 για να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να λειτουργεί, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Είναι θέμα τεχνικό, Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και θυμάμαι η Πορτογαλική Προεδρία η οποία είχε βοηθήσει να βρεθούν κάποιες λύσεις. Παρόλα αυτά τα νέα κράτη-μέλη δεν μπορούν σήμερα να προσχωρήσουν στο Σέγγεν. Χρειάζονται περισσότερα κονδύλια έτσι ώστε να υπάρξει η τεχνική υποδομή του ΣΥΣ 2 όπως χρηματοδοτήθηκε και η πρώτη φάση το ΣΥΣ 1. Χρηματοδότηση λοιπόν, γιατί όπως ξέρετε πρόκειται για κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογούμενων και θα πρέπει να δούμε αν οι επενδύσεις που έχουν γίνει έχουν γίνει με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να υποφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πιστεύω και εγώ ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί παρά να αυξήσει την ασφάλεια στην ε, Ευρώπη. Τώρα, το θέμα των καθυστερήσεων. 2001, 2002 μέχρι το 2007 το σύστημα θα έπρεπε να λειτουργεί. Έχουν περάσει 10 χρόνια σήμερα από το ξεκίνημα. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόση αβεβαιότητα και τόσοι αστάθμητοι παράγοντες που να επηρεάζουν ένα τέτοιο ε, σύστημα. Τεράστιες καθυστερήσεις και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι ποιος είναι ο λόγος, τι κρύπτεται όπισθεν. Μήπως κάποιοι οποίοι δεν θέλουν να προχωρήσει το σύστημα. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο και με το ΒΙΣ όπως έγινε και με το ΣΥΣ. Και πώς μπορούμε να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα. Ευχαριστώ πολύ και βάσει της διαδικασίας ΚΑΤΣΔΙ η κυρία Λουκάτσεβα θέλει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, ε, λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης και εφαρμογής του ΣΥΣ 2 Φοβάμαι ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν θα είναι έτοιμο ούτε το 2012 ούτε το 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να, κάνει, να προβεί σε κάποιες δοκιμές εάν αποδειχθεί, αν αποδειχθούν οι δοκιμές ανεπαρκείς, τι θα γίνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα αλλακτικό σχέδιο Τι θα γίνει με τις επενδύσεις που έχουν κάνει ορισμένα κράτη-μέλη αγοράζοντας εξοπλισμό για να εφαρμόσουν το νέο σύστημα ή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά, τα, αυτόν τον εξοπλισμό για να λειτουργήσουν το, παλιό σύστημα, το ΣΥΣ και όχι ένα και όχι το ΣΥΣ 2. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητάει το λόγο, γι' αυτό θα επανέλθω στην Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, κύριε Μπαρό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που, μου τέθηκαν, διότι για το ΒΙΣ, όπως σας είπα, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των δοκιμών που πρέπει να γίνουν μέχρι τις 11 Νοεμβρίου και για το SIS 2 ε, μιλάμε Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα του, των τεχνικών κριτηρίων που πρέπει να πληρωθούν ε, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Πράγματι, θα ήθελα να συμμετέχει άμεσα και ενεργά σε όλη τη διαδικασία ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα δύο μεγάλα σύστημα, σας θυμίζω, σχεδιάστηκαν από τα κράτη-μέλη για να ισχύει η ελευθερία κυκλοφορίας ε, μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης ασφάλειας όπως θύμισε ο κύριος Μπουζουτήλ για το ΒΙΣ. Θα ήθελα να πω στην κυρία Λάτφορντ, η οποία ως εισηγήτρια παρακολούθησε από κοντά αυτό το θέμα, το ΒΙΣ λοιπόν για το ΒΙΣ θα γίνουν οι δοκιμές μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, οι οποίες θα μας πούν εάν θα χρειαστεί να αλλάξουμε πορεία. Μέχρι στιγμής το σύστημα ΒΙΣ πιστεύουμε έχει ικανοποιητική αρχιτεκτονική. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά. Από τις δοκιμές λοιπόν που θα γίνουν τώρα θα διαπιστώσουμε κατά πόσο πρέπει να λύσουμε τη σύμβαση. Είναι όμως νωρίς να το πούμε αυτό ακόμα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ε, χρειαστεί να, να αναθεωρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Σας θυμίσω ωστόσο το 2005 το Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμόζεται με συντονισμένο και συνεπή τρόπο το βίσα από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό προβλέπεται ότι θα αρχίσει στην πρώτη περιοχή την ημερομηνία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν όλα τα κράτη-μέλη θα την έχουν ενημερώσει ότι προέβησε σε αναγκαίες νομικές και τεχνικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του ΒΙΣ σε αυτή την περιοχή. Το ΒΙΣ λοιπόν θα αρχίσει κανονικά να λειτουργεί στην πρώτη περιοχή που είναι η Βόρεια Αφρική που καλύπτει τις χώρες που αποτελούν το σημαντικότερο κίνδυνο στον τομέα της ασφάλειας και της λατρομετανάστευσης την ίδια ημερομηνία για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό με κάνει να πω ότι είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να εφαρμόσουν σε επιχειρησιακό επίπεδο το ΒΙΣ ότι θα ήταν πολύ δυσάρεστο αν το κεντρικό σύστημα αποδειχθεί ότι λειτουργεί ομαλά και λόγω καθυστερήσεων σε ορισμένα να υποχρεωθούμε να, παρατείνουμε ξανά τις προθεσμίες. η κυρία Λάτφοντ αναφέρθηκε στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε προχωρήσει αλλά ξέρω ότι έχει προβλεφθεί ότι το το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει δυνατότητα να συνδεθεί με το SIS 1 συν, το ενισχυμένο SIS συν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Για τους ετούντες θεωρήσεις ελπίζουμε ότι θα τηρήσουμε λίγο πολύ την προθεσμία που είχε οριστεί, διότι είναι πολύ σημαντικό για μας να αποφύγουμε το visa shopping στα προξενία, κάτι που υπάρχει κίνδυνος να συμβεί εάν καθυστερήσει υπερβολικά η λειτουργία του ΒΙΣ. Η κυρία Όσκα αναφέρθηκε στα βιομετρικά στοιχεία και ε, τον έλεγχο της πρόσβασης στο σύστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ο έλεγχος αυτός θα υπάγεται σε μια σειρά από σαφείς κανόνες. Η κυρία Έρνστ διαπίστωσε ότι είναι κατά του συστήματος και έρχομαι τώρα στον κύριο Κοέλο. Ο κύριος Κοέλο γνωρίζει πολύ καλά το SIS-2 και θα προσπαθήσω να του δώσω κάποιες απαντήσεις επιφυλασσόμενος να του δώσω και γραπτός τις υπόλοιπες απαντήσεις στις 7 ερωτήσεις του. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τις διαπραγματεύσεις, τις συμβατικές με τον ανάδοχό της, που οι διαπραγματεύσεις αυτές κάλυψαν δύο σκέλη. Τα συμπληρωματικά, ό,τι τα συμπληρωματικά που χρειάζονται για την ε, διεξαγωγή των δοκιμών, για την επίτευξη του τεχνικού ορόσημου. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία τέλη λίου και ο ανάδοχος ε, τότε είχε παρατηρήσει ότι υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές για το σύστημα που δυσκόλευαν πάρα πολύ την επίτευξη αυτού του πρώτου milestone. Παρ' όλα τα αυτά υπογράψαμε μία σύμβαση με τον ανάδοχο η οποία προβλέπει την ολοκλήρωση, την επίτευξη αυτού του milestone, του ορόσημου. Η περίοδος ανάλυσης και επισκευής μας επέτρεψε να δούμε, να διαπιστώσουμε ότι το ΣΥΣ 2 βασίζεται σε υγιείς βάσεις, αν και ε, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Και βρήκαμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τρόπους για τη βελτίωση του συστήματος. Κύριε Κοέγιο, και το λέω για όλους τους βουλευτές, Έχουμε ένα σχέδιο πάρα πολύ φιλόδοξο και δεν είναι εύκολο να, δούμε, να, να, μαντέψουμε το τι θα συμβεί. Εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον συνεταιρισμό, με το consortium Hewlett Packard Stereo, ε, αποζημιώσεις και πρόστιμα. πρόστιμα σε περίπτωση που δεν θα είναι λειτουργικό το σύστημα κατά το τέλος της σύμβασης όπως επίσης και για τις καθυστερήσεις για τα εσωτερικά τεστ του ΒΙΣ. Και τα δύο σχέδια έχουν, ε, διέπονται από το ίδιο συμβόλαιο. Αυτά τα πρόστιμα λοιπόν είναι πάνω κάτω 3,5 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα ε, συνεχίζουμε να μετράμε τα, τις καθυστερήσεις για το ΒΙΣ ενώ έχουμε σταματήσει με τα πρόστιμα του ΣΥΣ. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρξει εγκατάλειψη του σχεδίου, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστεί το κόστος. Ε, αισθάνομαι περίεργα απέναντι στο κοινοβούλιο αλλά σε αυτήν τη φάση κυρία Πρόεδρε καταλάβετε με δεν μπορώ να πω για το ΣΥΣ στις 11 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουμε κάποια αποτελέσματα και για το ΒΙΣ στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε το Milestone για να δούμε αν όντως είναι ένα σχέδιο που μπορεί να σταθεί Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να απαντήσω προκαταβολικά δυστυχώς. Το κοινοβούλιο πολύ ευχαρίστως να έρθει να, να, εξετάσει και αυτό το κόστος ε, ε, ελπίζω όπως και με το, με το Γαλιλαίο θα καταφέρω να σώσω αυτά τα δύο σχέδια που είναι πολύ αξιόλογα από τεχνολογικής πλευράς αλλά ακόμα δεν μπορώ να έχω τη βεβαιότητα από απόψε. Επίσης το Κοινοβούλιο έχει το καλωσόρισες για να μπορέσει να σμπρώξει λίγο τα κράτη-μέλη. Γιατί στο, οι καθυστερήσεις ε, του ΒΙΣ οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις ορισμένων κρατών μελών. Αυτό τα κυρία Πρόεδρε, ε, το ξέρω ότι δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά στο βαθμό που θα μου έρχονται και οι πληροφορίες είμαι έτοιμος και εγώ να απαντάω στα ερωτήματα των βουλευτών. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο για τις απαντήσεις που μας έδωσε και τελειώνοντας έχω τρεις προτάσεις ψηφίσματος οι οποίες θα περάσουν από ψηφοφορία την Πέμπτη. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι λίγη η σημερινή συνεδρίαση και η επόμενη θα είναι αύριο το πρωί με την ημερήσια διάταξη η οποία έχει δημοσιευθεί και στο έγγραφο της συνεδρίασης αλλά